Υπότιτλοι AUTHORWAVE Υπότιτλοι AUTHORWAVE Υπότιτλοι AUTHORWAVE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

Και εγώ δεν το είχα δει, δεν το είχα δει. Ακόμα να δει, δεν το είχα Του λέμε τα του λέμε τα δεύτερα, του λέμε τα δεύτερα. Εγώ δεν το είχα δει. Αυτό το οποίο να πει Ευχαριστώ.